Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε και πάλι, μετά από 18 χρόνια. zaszczyt i przyjemność dla Έχουμε την τιμή και χαρά να καλωσορίσουμε σήμερα μεταξύ μας τον πρόεδρο τη Δημοκρα... της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ανατολικού Τιμπόρου, θα θυμάστε την ομιλία του κυρίου Χωσέρα Μος Χόρτο πριν από 18 χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχε αναφερθεί στην ε, κατάσταση στον Ανατολικό Τιμόρ, το οποίο ακόμη τότε δεν ήταν ανεξάρτητο. Μόνο λίγοι ήταν εκείνοι οι θαραλέοι που τόλμησαν ε, να παρουσιάσουν οράματα τόσο τολμηρά όπως η ανεξαρτησία του Ανατολικού Τιμόρ. Ως δραστήριο μέλος της αντιπολίτευσης, ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έπεισε με την παρουσία του και τα επιχειρήματά του ως ο κύριος αγωνιστής για την ανεξαρτησία του Τιμόρ, του Ανατολικού Τιμόρ, με πέντε σημεία σε μια έκθεση που προέβλεπε και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και την ε, ε, εγκατάσταση διεθνών στρατευμάτων για την διαφύλαξη της ειρήνης και το, η διεξαγωγή του υποψηφίσματος για την ε, ανεξαρτησία. Ε, σχέδιο πέντε σημείων το οποίο αναγνώρισε και ενέχνε και η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996. Κύριε Χωσέ Ραμός Χόρτα και εσείς όπως και ο κύριος Ριμπέιρο ε, τιμηθήκατε με το βραβείο Νόμπελ της Ειρήνης. Στη συνέχεια ο κύριος Ραν Κουσμάο τιμήθηκε και εκείνος με τη σειρά του με το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στη συνέχεια διεξήχθη το δημοψήφισμα για τον Ανατολικό Τιμόρ, στο οποίο ε, εγκρίθηκε η ανεξαρτησία, ύστερα από την οποία ξεκίνησε μια δύσκολη περίοδο συμφιλίωσης στη χώρα, μέσα από την οποία θεσπίστηκαν αξιόπιστοι και δημοκρατικοί θεσμοί, η κοινωνία των πολιτών, μια πορεία μέσα, από την, μέσα στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στάθηκε πάντοτε αρρωγός στο Ανατολικό Τιμόρ και υποστήριξε πάντοτε τις προσπάθειες και του κυρίου Προέδρου αλλά και του Δημοκρατικού Κινήματος εν γέννη στη χώρα αυτή. Το 2002 ανέκτησε την πλήρη αναξαρτησία της η χώρα και πρέπει να σημειώσω ότι η εμπειρία του κυρίου Προέδρου Χωσέ Ραμός Χόρτα είναι πολύτιμη. Πρόκειται για έναν ε, ηγέτη ο οποίος ε, περιοδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο, προσφέρει την, τη μαρτυρία του και την εμπειρία του και σε χώρες που ακόμη δεινοπαθούν δίνει συμβουλές και αισιοδοξία ότι μπορούν να βρούνε το δημοκρατικό δρόμο και την ανεξαρτησία για τους πολίτες τους. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω τις παρατηρήσεις μου στα αγγλικά και μετά θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Μετά ξανά στα αγγλικά. Θα μπορούσα να σας μιλήσω σε πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες. Δεν θα το πράξω όμως, για να μην συγχυστώ και ο ίδιος θα περιστώ σε δύο αγγλικά και πορτογαλικά. Είμαι ευγνώμων για την τιμή αυτή που μου κάνετε να απευθυνθώ στο αξιοσέβαστο αυτό πολιτικό σώμα που αποτεί φόρο τιμής στην πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Ο θαυμασμός μου για την Ευρώπη και τους θεσμούς της είναι γνωστός. τον δρόμο που ακολουθήσατε για να γεφυρώσετε τις διαφορές σας και να οικοδομήσετε εταιρική σχέση, ευημερία καθώς και τα πιστεύω σας για το αλληλεγγύη μεταξύ λαών με οδήγησαν και εμένα που έχω λάβει τον Νόμπελ Ειρήνης το 2008 να ορίσω με τη σειρά μου την Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποψήφιο ε, για το Νόμπελ Ειρήνης. Γιατί η μόνη υπερδύναμη που υπάρχει αυτή τη στιγμή και απ' την άλλη οι οικονομικοί γίγαντες της Ασίας βρίσκουν την Ευρώπη στη μέση που μπορεί να και πρέπει να αποτελέσει γέφυρα που να τις συνδέσει σε μια νέα εταιρική σχέση ειρήνης και ευημερίας. Η Ευρώπη αυτή της συμπερίληψης αρχίζει από την όμορφη ακτή του Ατλαντικού μέχρι τις παρυφές της Παλαιάς Υπήρου όπου αρχίζει η Ασία. Τη στιγμή που σας μιλώ Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα δε τον πρόεδρό της, τον φίλο μας Ζουζέ Μανουέλ Δουράν Μπαρόζου, που στάθηκε αρρωγός σε όλο μας τον δρόμο του αγώνα για την ελευθερία και ως διπλωμάτης και ως πολιτικός στη χώρα του και ως Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας υπήρξε σοφός και πιστός φίλος του Ανατολικού Τιμόρ. Δεν θα ήταν όμως σωστό να μην ευχαριστήσω και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μερικά δυστυχώς απεβίωσαν, λόγω της ε, ανικές του γυράνσεως την οποία δεν μπορεί κανείς να αποφύγει και που από όλες τις πολιτικές παρατάξεις μας χορήγησαν ένα βήμα και μια φωνή που δεν μας έδινε κανείς άλλος. Παραδείγματος χάρη οι Πορτογάλοι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων που τη δεκαετία του 90 έδωσαν, χορήγησαν ένα τμήμα του μισθού των στον τωρινό μας πρωθυπουργό τον δόκτορα Ζαχαρία Κώστα που ήταν τότε εκπρόσωπος της αντίστασης στο Τιμόρ και Πορτογάλος Ευρωβουλευτής. Οκ, και τον υποστήριξαν όλοι οι Πορτογάλοι ευρωβουλευτές και αριστεροί και δεξιοί. Από εκεί επίσης για πρώτη φορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγήθηκε για πρώτη φορά τιμωρική ταυτότης. Έρχομαι λοιπόν εδώ μετά από τόσο καιρό με τεράστιο αίσθημα ευγνωμοσύνης προς όλους σας. Τώρα θα στραφώ προς την Πορτογαλική για να μιλήσω για το θέμα των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και πώς τους εφαρμόζουμε στη χώρα μου, καθώς και τι αναμένουμε από τη διεθνή κοινότητα για να μας βοηθήσει στην επίτευξή τους. Το τιμό ρολέστη δεν ήταν ανεξάρτητο το 2000. Και άρα πρόκειται για την πρώτη μας έκθεση για τους στόχους της χιλιετίας το 2004 όταν ε, δηλαδή είδαμε ποια ήταν τα, οι πρώτοι στόχοι που θα έπρεπε να επιτύχουμε. Στα τελευταία τρία χρόνια στο Ανατολικό Τιμόρ πραγματικά ζούμε μια ειρηνική περίοδο που διευκόλυνε την οικονομική ανάπτυξη πάνω από 2%, 12% ε, ετησίως. Ε, μειώθηκε η φτώχεια κατά 9% κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Περιορίστηκε η παιδική θνησιμότητα και η βρεφική θνησιμότητα κοινότητα, φτάνοντας μάλιστα στους στόχους που έχουν ε, καθιερωθεί, που έχουν θεσπιστεί για το 2015. Επίσης ε, η φίτηση στα σχολεία αυξήθηκε κατά, στο, και έφτασε στο 83% το 2009 και 2010. Ο αναλφαβητισμός των, ε, των ενηλίκων ανθρώπων έχει επίσης σχεδόν εκριζωθεί χάρη σε ένα κοινό πρόγραμμα ανάμεσα στο Ανατολικό Τιμόρ και την Κούβα. Ήδη προβλέπουμε την εκρίζωση του αναλφαβητισμού στο Ανατολικό Τιμόρ σε δύο με τρία χρόνια. Γύρω στο 30% του γενικού προπολογισμού του κράτους ε, χορηγείται αυτή τη στιγμή για την υγεία και την παιδεία. Αυτή η μεταστροφή συνέβη χάρη σε μια επιθετική δημόσια πολιτική επενδύσεων μέσω άμεσης ε, μεταφοράς χρημάτων για τους ε, ηλικιωμένους, τις χείρες, τους βετεράνους πολέμου, ώστε να μπορέσουν να επεκταθούν και σε περιοχές όπου ε, παλιότερα ήταν εγκαταλειμμένες, να βελτιωθεί η κατάσταση της γεωργίας ε, και η αυτονομία μας. Το στρατηγικό μας πρόγραμμα ε, προβλέπει μέχρι το 2030 το ότι θα εκριζωθεί η φτώχεια που ταλανίζει τη χώρα μας εδώ και αιώνες και ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια μεγάλη ευρύτατη μέση τάξη μέχρι το 2030. Σε σχέση με τα, τους πετρελαϊκούς μας πόρους, με ικανοποίηση μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η πρωτοβουλία διαφάνειας των εξωτερικών βιομηχανιών, δηλαδή Extractive Industries ε, και η πρωτοβουλία τους ε, μπόρεσε να αναφέρεται μάλιστα και στην αναφορά του 2010 ως τη τρίτη χώρα στην Ασία ε, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προσόδων από την εκμετάλλευση φυσικού αερίου και πετρελαίου. Γύρω στο 30% των βουλευτών στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο είναι γυναίκες στο εκτελεστικό στα Υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης και τα λοιπά, εκεί έχουμε υπουργού γυναίκες. Έχουμε ένα μόνιμο κοινοβούλιο νέων με 130 μέλη που μόλις εξελέγησαν από ολόκληρη τη χώρα οι νέοι που εξελέγησαν γι' αυτό το, το Κοινοβούλιο Νέων είναι ηλικίας μεταξύ 12 και 17 ετών. Ανέκαθεν ήταν επιθυμία μας να υπάρξει ισορροπία των φίλων στο Κοινοβούλιο των Νέων. Ήταν λοιπόν προσδοκία μας ε, αυτή, αλλά ξεπεράστηκε, γιατί το Κοινοβούλιο των Νέων αποτελείται κατά ε, από 68 βουλευτές θηλυκού γένους και 62 αρσενικού γένους. Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε υιοθετήσει ένα από τα πιο ανθρωπιστικά συντάγματα του κόσμου όπου η θανατική ποινή απαγορεύεται. και η μέγιστη ποινή κάθριξη είναι 25 έτη. Δεν υπάρχει ισόβια κάθριξη, δεν προβλέπεται. Επικυρώσαμε όλες τις βασικές διεθνείς συνθήκες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήδη παρουσιάσαμε δύο εκθέσεις για τις ε, συνθήκες αυτές στα αρμόδια όργανα και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας για όλους. Το Σύνταγμά μας αναγνωρίζει ότι υπερέχει το διεθνές δίκαιο των εθνικών νόμων. Δηλαδή, όλη μας η νομοθεσία θα πρέπει να συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα μιλήσω πάλι στα αγγλικά. Και θα απευθυνθώ τώρα, θα αναφερθώ τώρα στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Πολύ επιφανειακά βέβαια, λόγω και του περιορισμένου χρόνου που έχω στη θέση μου. Είναι δεδομένο ότι οι ισχυρές και οι ισχυρίες και πλούσιες χώρες έχουν συμβάλει στην επιδείνωση της κλιματικής και των περιβαλλοντικών, ε, του κλίματος και των περιβαλλοντικών συνθήκων κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα τελευταία 200 χρόνια έχουν οι μεγάλες αυτές και βιομηχανικές χώρες προσφέρει και μεγάλα ωφέλη στον κόσμο, έστω και αν δεν ήταν ισότιμη η κατανομή αυτών των ε, εκτιμάτων. Όμως εμείς στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν μπορούμε να κατηγορούμε για τα πάντα τους ε, πλούσιους και ισχυρούς. Δεν μπορούμε να τους κατηγορούμε για το κακό, για τα δεινά που υφίσταται ο πλανήτης. Πρέπει να ε, αναλάβουμε και εμείς το μέρος της ευθύνης που μας ανήκει για την καταστροφή των τροπικών δασών, την καταστροφή και ρήπανση των λιμνών, θαλασσών και ποταμών. Έχει λοιπόν και η Ασία, όπως και η Ευρώπη, η Αμερική, την ευθύνη της, το μερίδιο της ευθύνης ως προς την ανατροπή των, ε, ε της επιδείνωσης ε, των περιβαλλοντικών συνθήκων. Εκπροσωπούμε σχεδόν το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού. Έχουμε λοιπόν μερίδιο και στην κατανάλωση, η επιδείνωση ε, του επίπεδου των υδάτων, του περιβάλλοντος, των δασών. Χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερη ενέργεια, ενέργεια που παράγεται από τον πλανήτη Γη και όλο και περισσότερες είναι σχετικές χώρες οι οποίες ε, πέραν των ωκεανών και των θαλασσών αναζητούν ε, ενεργειακές πηγές ε, από άλλες υπήρους, ακόμη και από την Αφρική ή την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν το Ανατολικό Τιμόρ μαζί με τις Μαλδίβες δύο από τις μικρότερες δηλαδή χώρες της Ασίας, ενώσαμε τη φωνή μας για να ζητήσουμε μια κοινή ατζέντα, ένα κοινό πρόγραμμα της Ασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη, για την προστασία και την ανάκτηση του περιβάλλοντος, για την διαχείριση των εδαφών και των υδάτων, υγεία και εκπαίδευση για τους πάντες, για ε, ε, εκρίζωση της φτώχειας και του αναλφαβητισμού έκκληση προς τους ισχυρούς και προς τους πλούσιους. Οι πλούσιοι και οι ισχυροί θα πρέπει να διαρωτηθούν εάν έχουν υλοποιήσει τις μεγάλες προσχέσεις που έκαναν ενώπιον των τηλεοπτικών ε, φακών και αν έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της υπανάπτυξης και της φτώχειας. Κατηγορούνται η, οι ανε, αναπτυσσόμενες χώρες για την ε, μη εξασφάλιση των στόχων της ανάπτυξης υπέρ των λαών μας. Λέγεται ότι δεν αξιοποιήσαμε δηλαδή τα χρήματα που λάβαμε ως ε, ενίσχυση, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και τι έχει στην πραγματικότητα συμβεί. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σαφές ε, αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των απλών ανθρώπων. Στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη ή την Ιαπωνία ο απλός άνθρωπος έχει αίσθημα αλληλεγγύης απέναντι στον συνάνθρωπό του στις πιο φτωχές περιοχές του κόσμου. Αλλά ταυτόχρονα οι χορηγοί θα πρέπει να καθοδηγήσουν τα κονδύλια κατά τρόπο ώστε να μην είναι επαναληπτική, γραφειοκρατική, βαριά, περιττή ή και δαπανηρή ακόμα η διαδικασία που τα οδηγεί σε εκτέλεση. Οι θα πρέπει να επενδύουν περισσότερο την κάθε δεκάρα την οποία υποσχέδεται ότι θα προσφέρουν στη γεωργία, την, ε, τα καθαρά ύδατα και εδάφη, τις οδικές, εξωτικούς άξονες, την υγεία και την εκπαίδευση, την ενίσχυση των εθνικών και δημοκρατικών θεσμών την υποστήριξη των δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών. Και γι' αυτό το στόχο θα πρέπει να προσφέρουν οι δωρητές, οι χορηγοί, πιο τομεακά οργανωμένες ενισχύσεις που θα στοχεύουν ακριβώς στην ενίσχυση, στην ε, κάλυψη των αναγκών των λαών. Μόνο έτσι και πρέπει να σημειώσουμε ότι ελάχιστες είναι οι πλούσιες χώρες οι οποίες ε, ικανοποίησαν το στόχο του 0,7% του μεικτού ΑΕΠ σε, ως αναπτυξιακό στόχο και ενώ ταυτόχρονα γενναιόδορες υποσχέσεις που δόθηκαν κάτω από το φως των προβολέων μαζί με ηθοποιούς του Χόλιγουτ και αστέρες της ροκ μουσικής λησμονήθηκαν όπως γρήγορα καταραίουν και τα σκηνικά στο Χόλιγουτ όπως γρήγορα σβήνουν και οι προβολείς της δημοσιότητας. Έτσι λοιπόν είδαμε δεκάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων να ε, βρίσκονται εύκολα και γρήγορα για να προστατευθούν και να διασωθούν από την κατάρρευση ε, είτε τράπεζες, είτε επιχειρήσεις, είτε βιομηχανίες που πολλές φορές είχαν καταχραστεί και δημόσιο χρήμα είχαν κάνει ψευδείς δηλώσεις. Ή εκατομμύρια πριν χορηγούνται σε ε, διευθυντικά στελέχη των μεγάλων ομήλων που κατά τα άλλα κατηγορούνται για οικονομικές ατασταλίες. Όμως τα ποσά αυτά που χρειάζονται τα αναπτυσσόμενα κράτη βρίσκονται πάντοτε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Πάντοτε αντιμετωπίζουν πολλές αντιδράσεις, τα αιτήματα για χρηματοδότηση των φτωχότερων κρατών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι σοφός και τίμιος, έντιμος τρόπος για υποστήριξη των φτωχότερων χωρών που υποφέρουν από την οικονομική κατάρρευση και την κρίση θα ήταν η διαγραφή των χρεών των λιγότερων επιτυγμένων κρατών και των φτωχών κρατών και η αναδιάρθρωση των χρεών, των χρεωμένων κρατών που έχουν τεράστιες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις όπως αστάθεια, κλιματική αλλαγή, εξτρεμιστικές τάσει και οργανώσει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιε χώρε όπω το Ανατολική Ασία, αλλά και στην περιοχή των μεγάλων λιμνών τη Αφρική. Το Τιμόρ Λέστε, το Ανατολικό Τιμόρ, έχει την τύχη να μην έχει ούτε ε, μίας δεκάρας εξωτερικό χρέος. Άρα η έκκληση που σας απευθύνουμε δεν υποκινείται από εγωιστική η σκοπιμότητα. Και αν κοιτάξετε το Economist, το Yearbook, δηλαδή την επιτηρίδα για το 2010 που εκδίδει το περιοδικό Economist θα δείτε ότι σε σχέση με το ΑΕΠ του το Ανατολικό Τιμόρ έχει το μεγαλύτερο πλεόνασμα κατέτος χωρίς ούτε, ένα, ούτε μία δεκάρα σε εξωτερικό χρέος παρόλα αυτά εμείς στασόμεθα αλληλέγγυοι με τα κράτη εκείνα τα οποία ε, ε, γονατίζουν κάτω από το βάρος του εξωτερικού τους χρέους, είναι σε αδυναμία να το εξυπηρετήσουν και οδηγούν σε απελπισία οι συνθήκε αυτές εκατοντάδες εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον κόσμο. Εάν μπορούμε λοιπόν να βρούμε μερικά δισεκατομμύρια δολάρια από τη μια μέρα στην άλλη για να σώσουμε κάποια τράπεζα από την πτώχευση ή κάποια ασφαλιστική εταιρεία από την κατάρρευση, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν γιατί είναι ηθική υποχρέωση πολιτική σοφία και ευφυΐα να βρεθούν πολύ λιγότερα μάλιστα ποσά για να στηριχθούν οι χώρες αυτές, να σβηστεί το, το χρέος τους ή να, δοθούν, να δοθεί μια χείρα ε, βοηθείας προς τους πιο φτωχούς στον κόσμο. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Ομιλώ σήμερα εδώ με βαθύτατο αίσθημα ευγνωμοσύνης προς εσάς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους Ευρωπαίους ηγέτες, προς όλους τους αναπτυξιακούς μας εταίρους και ταυτόχρονα με ταπεινοφροσύνη αναγνωρίζω και τα σφάλματά μας και τα όρια των δυνατοτήτων μας. Εμείς, στον Ανατολικό Τιμόρ και στο, στο μεγαλύτερο μέρος του αναπτυσσομένου κόσμου, θα πρέπει να αποφύγουμε την ανατροπή ρόλων. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κηρύγματα στην Δύση, όταν σταματάει η Δύση να κάνει κηρύγματα σε εμά για το πώς θα σώσουμε τον κόσμο. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα στον καθρέφτη και να ρωτήσουμε τη συνείδησή μας τι κάναμε, τι έχουμε πράξει για να απαλλάξουμε τα εκατοντάδες των εκατομμυρίων των συμπολιτών μα από τι ακραίε συνθήκε φτώχειας και εξαθλίωση. Μπορούμε να πράξουμε πολλά, μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε περισσότερο και στον Ανατολικό Τιμόρ αλλά και στα άλλα κράτη. Έχουμε πραγματοποιήσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Οχτώ χρόνια έχει μόλι ανεξαρτησία η πατρίδα μου. Κάποια από τα αριθμητικά στοιχεία σα τα έδωσα. Όμω υπάρχουν πολλοί άλλοι τομεί επιτεύγματα τα οποία δεν μπορούμε ποσοτικά να προσμετρήσουμε, δεν μπορούν να υπολογιστούν σε αριθμούς, αλλά έχουν επίσης ε, ύψιστη σημασία. Φερρυπίν, μπορέσαμε να θεραπεύσουμε τις πληγές, τις κοινωνικές πληγές, να συμφιλιώσουμε διχασμένες κοινωνίες, να ε, καταρρύψουμε τα τείχη μεταξύ ημών και της Ινδονησίας, με την οποία μας ενώνει μια τραγική ιστορία 24 ετής. Σήμερα η Ινδονησία και το Ανατολικό Τιμόρ έχουν τις βέλτιστες δυνατές σχέσεις γειτονίας. Μπορέσαμε να οικοδομήσουμε γέφυρες με ολόκληρη την περιοχή μας. Έχουμε διπλωματικές σχέσεις με άνω των 100 κρατών. Μη προσμετρούμενα επιτεύγματα, όπως έλεγα, δεν μπορούν να υπολογιστούν σε στατιστικά στοιχεία. Ο λαός μας, παρά τα δεινά των 24 ετών και της κυριαρχίας, της ξένης κυριαρχίας, δεν τρέφει συναισθήματα αντεκδίκησης εναντί ουδενός. Αυτή είναι η πεποίθησή μας, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Είμαστε αποφασισμένοι να ανέλθουμε στο ύψος των προσδοκιών των συμπολιτών μας και να εργαστούμε σκληρά για ένα μέλλον ευημερία και ειρήνης. Και ελπίζω ο φιλεύθυνος Θεός να μας στηρίξει και να σας ευλογεί όλους. Ευχαριστώ πολύ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από 18 χρόνια ως ηγέτης της αντιπολίτευσης του Ανατολικού Τιμόρ με μέγα και μέγα όραμα Σήμερα ως πρόεδρος του ελεύθερου και δημοκρατικού ανεξάρτητου τιμόρ της χώρας σας, ε, ε, συγχαρητήρια σε εσάς κύριε Πρόεδρε και ό,τι καλύτερο εύχομαι για εσάς και για τη χώρα σας και το λαό σας. Σας ευχαριστώ.